Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα πρακτικά της συνεδρίασης στις 25 και 26 ε, Μαΐου είναι διαθέσιμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιρρήσεις.